Dear Κυρίες και κύριοι, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ, καθίστε. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Θα σας τα πω στα γερμανικά. Καλημέρα. Σας εύχομαι. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Έχετε την ημερήσια διάταξη προς Σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερη η συνεδρίασή μας ε, στις 11 η ώρα περίπου. Θα ε, έρθει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας ε, στο πλαίσιο του Gender Mainstreaming Network. Έχετε την ημερήσια διάταξη μπροστά σας και θα ήθελα να ξεκινήσω ακριβώς από την ημερήσια διάταξη. Σήμερα προβλεπόταν ε, διαρθωτικός διάλογος με την Επίτροπο Έλενα Ντάλη. Δυστυχώς έπρεπε να κυρώσει την ε, συζήτηση αυτή και γι' αυτό ε, έχουμε προγραμματίσει τις 26 Μαρτίου να την προσκαλέσουμε. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Και έτσι φτάνω στις ε, ανακοινώσεις ε, της Προέδρου. Έχετε το πρόγραμμα μπροστά σας. Όπως σας είπα, θα έρθει ο Ντάβιτ Σασόλη. Ε, οι ώρες που δίνονται είναι ενδεικτικές. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να προλάβουμε. Μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ε, στη συνεδρίαση της 26ης ε, Ιανουαρίου οι συντονιστές ε, αποφάσισαν ο προϋπολογισμός και η απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Δύο Φύλων να πάνε στην ε, Επιτροπή ε, και επίσης έχουμε ε, το θέμα της φροντίδας των παιδιών και προβλέπεται η σχετική συνεργασία επιπλέον. Άδεια για ακρόαση στις 28 Μαΐου 2020 με θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ισότητα των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγικές προτεραιότητες. Και Έχουμε διακοινοβουλευτική συνάντηση στο πλαίσιο της ε, διεθνού ημέρας ε, για την εξάλληψη της βία ει βάρος των γυναικών τον Νοέμβριο του 2020. Επιπλέον, ε, το πρωί της 26ης Μαρτίου και το βράδυ της 6ης Ιουλίου στο Στρασβούργο θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση. Θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας ε, την, το, το τροποποιημένο ημερολόγιο και έτσι φτάνουμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης, ε, τις ψηφοφορίες ψηφοφορίες σχετικά με την έκθεση για τα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2018-2019 και έχουμε ε, εισηγήτρια την Σαμίρα Ραφαέλα. Ελπίζω όλοι να έχετε τις κάρτες σας ε, μαζί σας. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε από την τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ,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 αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά,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 73 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προχωράμε στην τροπολογία 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, αλλά θα ήθελα να το επαληθεύσουμε. Δεύτερο τμήμα της 103. Μία ψήφος λείπει. Ωραία. Λήξη της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. 103 το τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104, wer 104 υπέρ, κατά, mm. αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108, υπέρ, κατά, θα ήθελα να επαληθεύσουμε την 106, διότι ναι, έγινε κάποιο μπέρδεμα η ηλεκτρονική επαλήθευση της 106. Äh, äh, so, jetzt haben alle abgestimmt. So. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας λοιπόν. 12 ε, υπέρ, 17 κατά, 4 αποχές. Απορρίπτεται. 43 το δεύτερο τμήμα. Μου λένε μόλις ότι δεν ψηφίσαμε την 106 και ίσως γι' αυτό ε, έγινε το μπέρδεμα. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 106 σε δύο τμήματα. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, 106 υπέρ. 106, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106, το δεύτερο τμήμα υπέρ. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Την 108 την ψηφίσαμε ήδη, πάμε στην 43, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. 43, το δεύτερο τμήμα. Λήξη της ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 9 αποχές. Ε, είναι σαφές το αποτέλεσμα. Λυπάμαι που δεν το είδα. Τροπολογία 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και φτάνουμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τρία των αιτιολογικών σκέψεων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεν φαίνεται πολύ καλά. Θα ήθελα ε, να το επαληθεύσουμε παρότι μάλλον ήταν σχετικά ξεκάθαρο. Σας παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας. Έναρξη της ψηφοφορίας λοιπόν. Λίγο ακόμα. Μην, κουράζεστε ακόμη. Ένας λείπει. Ωραία. Λήξη της ψηφοφορίας. 23 ε, υπέρ, 17 κατά. <clears throat> Ήταν σαφές, ε, τα χέρια σας δεν έβλεπα. Προχωράμε στην επόμενη συμβαστική τροπολογία, την υπαριθμόν 5, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33, υπέρ. Κατά, Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές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 Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή ψηφοφορία. Παρακαλώ όσους εγκαταλείπουν την αίθουσα να το κάνουν αυτό όσο γίνεται πιο ήσυχα.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 Συνάδελφοι, προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, που είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021, το τμήμα 3. Συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο Ρομπέρτ Μπιετρών, στον οποίο θα, ήθελα να του δώσω το λόγο, αλλά δεν μπορώ διότι δεν είναι παρόν. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Τρεπμάτιτς, Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους του συναδέλφου Ρόμπερτ Μπιέντρον θα διαβάσω τη δήλωσή του. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να παραβρεθώ στη συνεδρίαση. Ω εισηγητή γνωμοδότη για τον προπολογισμό του 2021, ήθελα να πω το εξή. Παρόλο που οι γυναίκε είναι το ίμιση τη ανθρωπότητα, υφίστανται διακρίσει σε κάθε τομέα τη ζωή. Ακόμη και στι πιο ανεπτυγμένε χώρε μέλη. Ω εκ τούτου θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η συνεκτίμηση τη διάσταση του φύλου στον προπολογισμό να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα τη δημοσιονομική διαδικασία σε όλε τι φάσει και σε όλε τι δημοσιονομικέ γραμμέ. Επίση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, δαψιλή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που στηρίζουν την οικονομική ανεξαρτησία και γενικώ ανεξαρτησία των γυναικών. Θα πρέπει οι δημοσιονομικέ δαπάνε να προωθούν την ισότητα των φύλων και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομα και καλά μας τα είπανε. Δίνω τώρα το λόγο στις σκιώδεις εισηγήτριες. Ποια θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ. Εκ μέρους ε, των Πρασίνων η EFA θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπιέντρον για την προσπάθειά του και το συνεργάσιμο πνεύμα που επικράτησε στις ε, Επιτροπές. Για πρώτη φορά ο εισηγητή του Γενικού Προπολογισμού κάλεσε και τι άλλε επιτροπέ να καταθέσουν γνωμοδοτήσει για τι κατευθυντήριε γραμμέ για τον προπολογισμό. Και εκτιμούμε ιδιαίτερω αυτό το άνοιγμα και αυτό το βήμα εκ μέρου του Γενικού Εισηγητού. Είναι μεγάλη ευκαιρία για την Επιτροπή Γυναικών να προωθήσει τι προτεραιότητέ τη για τι κατευθυντήριε γραμμέ του προπολογισμού του 2021, γιατί ο προπολογισμό αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων μα. Και η κατανομή των πόρων είναι θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και για τα ζητήματα των γυναικών. Συμφωνούμε με το σχέδιο γνωμοδότηση του κυρίου Μπιέντρον. Θα θέλαμε όμως παρόλα αυτά να προσθέσουμε κάποια σημεία και αυτό θα το κάνουμε με τις τροπολογίες μας για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που μας δίνει η γνωμοδότηση. Καταρχήν, θα πρέπει να αναφέρουμε ρητά τη συνεκτίμηση τη διάσταση του φύλου στι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν κάνει ο εισηγητή στην γνωμοδότηση και θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτό το κενό. Γιατί η συνεκτίμηση του φίλου θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε όλες τις φάσεις του κύκλου πολιτικής. Επίσης, η συμπερίληψη του φίλου στον προϋπολογισμό. Και ευχαριστώ τον ε, Ρόμπερτ Μπιέτρο για τις προσπάθειες που κάνει να συνεκτιμηθεί, να ενσωματωθεί η διάσταση του φίλου στον προϋπολογισμό και να ληφθεί υπόψη την κατανομή των πόρων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή Γυναικών. Λυπούμαστε ιδιαιτέρως που στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ ή στα ελληνικά, δεν ε, περιλαμβάνεται ε, η δυνατότητα ενσωμάτωση του φύλου, η προώθηση της ενσωμάτωσης του φύλου. Αυτό θα θέλαμε να το επισημάνουμε στην γνωμοδότησή μας. Επίσης, να τονίσουμε τη σημασία που έχουν τα διαρθρωτικά ταμεία για τις γυναίκες. Θα θέλαμε να αυξήσουμε τα κονδύλια για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση και για μικρές ΜΚΟ, για ακτιβίστες ανθρωπίνων δικαιωμάτων γυναίκες ε, και για τις γυναίκες που προασπίζουν ε, τα δικαιώματα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, καθώς και τα κονδύλια του Μηχανισμού Γειτονία και Αναπτυξιακή Συνεργασία. Επίση, για το νέο, το νέο Ταμείο για το Άσυλο και την εσωμάτωση θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ενδοοικογενειακή βία και να ε, διευκολύνουμε την πρόσβαση στα δικαιώματα σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Σας ευχαριστώ θερμά. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο από τους κοιόδες συζητητές, από ό,τι βλέπω όχι ούτε ο κ. Μάτης θέλει να προσθέσει κάτι. Έτσι ολοκληρώσαμε πολύ σύντομα το θέμα αυτό. Τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 20 ε, ε, Φεβρουαρίου στις 5 ε, το απόγευμα. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι 10 και 39. Θα κάνουμε λοιπόν ε, ένα μικρό διάλειμμα, διότι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης ε, των δύο φύλων ε, και στις 11 η ώρα θα έρθουν οι βουλευτές από τις άλλες επιτροπές. Στις 11 λοιπόν θα ξεκινήσουμε. με ένα σύντομο διάλειμμα για καφέ λοιπόν. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση μέχρι τις 11.